που πρόκειται για την κοινή συζήτηση σχετικά με την φάρμακοεπαγρύπνηση με την έκθεση της κυρίας Λίντα Μακέβαν αναφορικά με την φάρμακοεπαγρύπνηση σε φάρμακα ανθρώπινης χρήσης καθώς επίσης και την έκθεση της κυρίας Μακάβεν πάλι για την φάρμακοεπαγρύπνηση τροποποίηση της οδηγίας 2001 ε, 83. Ο κύριος Επίτροπος ε, βρίσκεται στη θέση του, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσως ε, και τον λόγο έχει η κυρία Μακάβανο στη Thank you, Mr. President. I'm sure... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι βεβαία ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ κάποια στιγμή έχουμε πάρει ή συνεχίζουμε να παίρνουμε φαρμακευτικά προϊόντα. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα της ασφάλειας αυτών των φαρμακευτικών προϊόντων και την προηγούμενη εβδομάδα μια συνεδρίαση ειδικών που ασχολήθηκε με την αυτή νομοθεσία άκουσε για άλλη μια φορά ότι το 2010 σημειώνει την 50η επέτειο της θελιδομίδης. Θα θυμάστε, όπω θυμάμαι και εγώ και οποιοδήποτε άλλο στην ηλικία μου, τι σημαίνει θελιδομίδη, τι εικόνε των παιδιών εκείνων που γεννιόντουσαν χωρί άκρα. Α διδαχθούμε λοιπόν από την εμπειρία αυτή οι κυβερνήσεις ε, στη διάρκεια αυτών των 50 ετών ανέπτυξαν συστήματα φαρμακοεπαχρύπνησης γιατί απεδείχθη ότι οι κλινικές δοκιμές και μόνες δεν αρκούν για να είμαστε βέβαιοι ότι ένα φάρμακο το οποίο διατίθεται στην αγορά για κατανάλωση από τον άνθρωπο δεν θα έχει κάποιες παρενέργειες. Έγιναν λοιπόν σημαντικέ πρόοδοι και την προηγούμενη εβδομάδα σε εκείνη τη συνεδρίαση ε, ενημέρωσαν οι ειδικοί ότι χάρη στην, ε, ε, στις προόδους που έχει πετύχει μέχρι τώρα η επιστήμη, μερικές μόνο τον αριθμό ε, υποθέσεις παιδιών που γεννήθηκαν με ελλειπή μέλη θα αρκούσαν για να βγει εθαλιδομίδη από την αγορά. Όμως χρειάστηκαν κάποιες χιλιάδες παιδιά να γεννηθούν την εποχή εκείνη. Τώρα λοιπόν έχουμε προχωρήσει. Έχουμε και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία στο Λονδίνο που ασχολείται με τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί γιατί 500 εκατομμύρια άνθρωποι είναι ένα μία βάση γνώσης που μας επιτρέπει πολύ πιο ευχερός να ανοιχνεύσουμε παρενέργειες από ότι εάν είχαμε μόνο τον πληθυσμό ενός κράτους μέλους. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ήταν εκείνη που μας έχει επιτρέψει να προοδεύσουμε, να προχωρήσουμε και τα πρακτικά μέσα όπως η, βάση φαρμακοεπαχρύπνησης που είναι η μεγαλύτερη βάση φαρμακοεπαχρύπνησης στον κόσμο μας επιτρέπει εγκαίρως ε, να εντοπίζουμε παρενέργειες. Χρειάζεται όμως περαιτέρω από το 1960 είδαμε άλλα προβλήματα από φάρμακο όπως το Βίοξ ή το Βάντια, ένα φάρμακο που δινόταν για τον διαβήτη. Οι βουλευτές, όπως και το Συμβούλιο, έχουν προχωρήσει στην πρώτη ανάγνωση στη διαπραγμάτευση μιας πολύ καλής δέσμης μέτρων που θα ψηφιστεί αύριο και που πιστεύω θα βελτιώσει σημαντικά τη φαρμακοεπαχρύπνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κύριες ε, Αλλαγέ λοιπόν είναι το ζήτημα τη ΠΡΑΚ, δηλαδή τη Επιτροπή για την Εκτίμηση τη Επικινδυνότητα στο πλαίσιο τη φαρμακοεπαγρύπνηση, που είναι η ουσία τη υπόθεση, δηλαδή η ε, διερεύνηση της ασφάλειας των φαρμάκων από ειδικού, όχι μόνο κυβερνητικού, αλλά και με συμμετοχή και επαγγελματιών του τομέα της υγείας και ασθενών των ίδιων. Επίσης, θα έχουμε την άμεση αναφορά από ασθενείς στις εθνικές αρχές προβλημάτων. Και μάλιστα καλούμε τους ασθενείς ή ε, όσους χρησιμοποιούν τα φάρμακα να ενημερώνουν αμέσως για παρενέργειες που εντοπίζουν. Ε, για τα νέα προϊόντα επίσης ε, γνωρίζει ένας ειδικό στον τομέα της υγείας όταν χορηγεί ένα νέο φάρμακο ότι πρέπει να επαγρυπνεί ε, για την ε, ενδεχόμενη εμφάνιση παρενεργειών, πράγμα το οποίο όμω δεν γνωρίζει ο ίδιο ο ασθενή και γι' αυτό ενημερώνεται καλύτερα ο ασθενή. Η προσέγγιση η μονοθυριδική όπου και η ενημέρωση για τον ασθενή και η ε, ε, συμμετοχή του ειδικού του επαγγελματία του τομέα υγείας. Όλα αυτά παίρνουν μέσα από ένα σύστημα μόνο ενιαίο, χωρίς επικάλυψη, χωρίς απώλεια χρόνου όπως είχαμε μέχρι τώρα, αλλαγές μεγάλες τις οποίες ε, κύριε Πρόεδρε εγώ κρίνω ως πολύ χρήσιμες. Θα βελτιώσουν σημαντικά τη φαρμακοεπαγρύπνηση ως σύστημα στην Ευρώπη και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους εκείνους, όλους όσους μας, μας βοήθησαν ε, στην βελτίωση τη φαρμακοεπαγρύπνηση, στους ειδικού συναδέλφου, στην Ισπανική Προεδρία στο Συμβουλίο, τον την κυρία Μοντέρο και την ομάδα της που είναι εδώ παρούσα σήμερα. Εξαίρετη δουλειά έχετε κάνει. Την ε, γραμματεία του Κοινοβουλίου, τους δικούς μας βοηθούς από την ομάδα μας όλους όσοι μελέτησαν τα πράγματα και τα... Ε, μας έδωσαν τις εξηγήσεις τους και την ερμηνεία τους με απλό τρόπο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, όλους έξω από το Κοινοβούλιο τους ενδιαφερομένους, εκπροσώπους ιατρών, ιατρικού προσωπικού, ε, εργαζομένους στον τομέα υγείας, ακόμη και ασθενών που μας ενημέρωσαν, μας έδωσαν στοιχεία και μας βοήθησαν στην υπόθεση αυτή. Τώρα ήρθε η ώρα να θέσουμε σε εφαρμογή ένα πολύ καλό κομμάτι νομοθετικού έργου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μακάβαν. Το, το λόγο έχει εκ μέρους της Επιτροπής ο κύριος Ταγιάννη. Ευχαριστώ πρόεδρα, Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο Επίτροπος Νταλή λυπάται που δεν μπορεί να παραστεί σήμερα το απόγευμα να ασχοληθεί με το ζήτημα και παρακαλεί να τον συγχωρέσετε. Εν τόσο έχω την χαρά να τον εκπροσωπώ για την έγκριση σε πρώτη ανάγνωση το, σχετικά με το ζήτημα της φαρμακοπαγρύπησης. Να δράξω την ευκαιρία λοιπόν προκειμένου να ευχαριστήσω όλους όσοι δούλεψαν για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Ιδιαίτερα την εισηγήτρια, τους συνεισηγητές, τους εισηγητέ, αλλά ιδιαίτερα την κυρία Μακάβαν, εισηγήτρια για το θέμα επί της ουσίας. Τώρα, χάρη στην πρόταση που θα πέρασει αύριο από το Κοινοβουλίο σα, ε, οι πολίτε θα είναι καλύτερα προστατευμένοι. Το σύστημα λοιπόν εισόδημα καβίβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχυθεί και θα εξυγχρονιστεί όχι μόνο για να προστατεύσει την δημόσια υγεία, αλλά θα διασφαλίσει και την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να ορθολογικεύσει τις διαδικασίες που σήμερα ισχύουν. Εξάλλου, η νομοθεσία θα αυξήσει την διαφάνεια και την συμμετοχή των ασθενών στον τομέα τη φαρμακοεπαγρύπνησης. Τέλο με την Επιστημονική Επιτροπή σε ζητήματα φαρμακοεπαγρύπνησης που συστάθηκε στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων θα υπάρχει πρόσβαση στην επιστημονική γνώση, την πλέον προκεχωρημένη για να βελτιωθεί η ασφάλεια των φαρμάκων και να προβλεφθούν μέτρα για τη μείωση των κινδύνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απόλυτα ικανοποιημένη που μια κοινή θέση μπόρεσε να προκύψει ανάμεσα στα τα εμπλεκόμενα μέρη πριν από τις διακοπές των πριν τερινές διακοπές. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό οι τροπολογίες που ε- έχει προταθεί προκειμένου να, ε, ε, να εκλεγεί ο, ο διευθυντής της ε, Τροπής ε, Φαρμάκων αντικαταστάθηκε από το εξή. Δηλαδή, με βάση τι αποφάσει του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σχετικά με το διευθυντή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων, η Κομισιόν θέλει να μην καθυστερήσει περαιτέρω αυτή η πρόταση και γι' αυτό δεσμεύεται να δημοσιεύσει την προκήρυξη προκειμένου να προσληφθεί ο ε, αρμόδιο διευθυντή στη θέση Α15 αντί για τη θέση Α14. Η Κομισιόν δεσμεύεται να συζητήσει το θέμα σε οριζόντιο επίπεδο σχετικά με τον ρόλο των υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο τη ομάδα εργασία τη Διόργανική που ασχολείται με το θέμα των υπηρεσιών. Ε, η εξέταση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει στο πλαίσιο τη διοργανική συνεργασία. Αν καταλήξουμε ότι η διευθυντή θα πρέπει να έχει διαφορετικό βαθμό. Αυτό θα ληφθεί υπόψη στι ε, περαιτέρω δημοσιεύσει για την προκήρυξη. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε την σα. Ολοκληρώσα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε. για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μηχανία Έρευνας και Ενέργειας το λόγο έχει για δύο λεπτά η κυρία Τιβάζη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα χρειαστώ ένα λεπτό και θα ξαναπάρω το λόγο ένα λεπτό αργότερα. Εδώ παρεμβαίνω συγητή για γνωμοδότηση της Επιτροπής Ήτρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Μακάβεν για την έκθεσή της και θα ήθελα να πω επίσης ότι για την υπόθεση αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των ασθενών και καλύτερη ενημέρωση, αλλά να καταπολεμήσουμε και την παρέμβαση της φαρμακοβιομηχανίας, η οποία ήθελε να, ε, έχει, να συγκεντρώνει πληροφορίες για τις παρενέργειες και να τις ερμηνεύει Επίσης, στα πλαίσια της ΣΥΤΡΕ, σε ό,τι αφορά το, τη συλλογή, εξασφαλίσαμε ότι οι ιατροί και οι ασθενείς θα ενημερώνουν για τις παρενέργειες στις εθνικές αρχές σε ό,τι αφορά την ανάλυση και την ερμηνεία αυτών των παρενεργειών, αυτό υπάγεται στην ευθύνη των κρατών μελών. Εκεί να καλούνται να παρακολουθούν και να υποπτεύουν τις παρενέργειες των ε, φαρμάκων. Οι Σουηδικές Εθνικές Αρχές συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στην αρκοληψία. Ενώ, ενώ μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε αυτές τις παρενέργειες αυτού του εμβολίου. Είναι λοιπόν σημαντικό. Εκεί που απογοητεύομαι ωστόσο είναι ότι εξασφαλίσαμε την οικονομική ανεξαρτησία των ε, εθνικών αρχών. Για τον έλεγχο υπήρξαν ουσιαστικές προόδεις σχετικά με την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης που είναι κάτι το χωριστό από την Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση και ελπίζω ότι η ενημέρωση για τον ασθενών θα είναι πληρέστερη στο ε, φύλλο χρήσης και στα ευρύτερα θέματα της φαρμακοεπαγρύπνησης. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της Επιτροπής Προστασίας ε, του Πολίτη, ο κύριος Τούρμες έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα λεπτό έχω ή δύο. Ένα. Α, τότε θα πρέπει να είμαι και πιο γρήγορος. Ε. Τα φάρμακα είναι βεβαίως μια επιχείρηση αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ και γι' αυτό το λόγο σκέφτηκαν και οι πιέσει των λόμπι της φαρμακοβιομηχανίας. Στην Επιτροπή των Οικονομικών της Ιστορικής Αγοράς τη εσωτερική αγορά, αυτό που καταφέραμε και τη προσθέσει του καταναλωτή, αυτό που καταφέραμε ήταν να ε, διατηρήσουμε ανοιχτό το φάσμα των θεμάτων που αφορούν την εσωτερική αγορά, όπω επισημάνθηκε και νωρίτερα, ε, με, τις, με την ταυτόχρονη παρακολούθηση της ε, παρακολούθησης των παρενεργειών των φαρμάκων και ταυτόχρονα να αποτρέψουμε τις πιέσεις της φαρμακοβιομηχανίας και, την, και να εξασφαλίσουμε την ενημέρωση του ασθενή με ε, επαρκή στοιχεία και όχι συνοπτικά. Δυστυχώ όμω βλέπω ότι από την έκθεσή μου δεν έγινε δεκτή μια ιδέα που θεωρούσα πολύ χρήσιμη, δηλαδή την παρακολούθηση τη θεραπευτική προσθέμενη αξία ορισμένων φαρμάκων, γιατί βλέπουμε τώρα ότι έχουν αναπτύξει κάποιες μεγάλες εταιρείε ε, μια νέα στρατηγική. Όταν λίγο πολύ λίγη η προστασία του, της μηχανικής διοκτησίας για ένα φάρμακο, το ε, μετατρέπουν κατά ορισμένα μόνο μόρια ή μικρομόρια και έτσι διατηρούν την προστασία του, χωρίς όμως αυτό να προσθέτει τίποτε σε σχέση με το ήδη φυστάμενο φάρμακο. Παραμένει δηλαδή το φάρμακο αυτό ακριβό γιατί είναι προστατευόμενο ε, προστατευόμενη ευρεσιτεχνία, αλλά δεν έχει τίποτα να προσφέρει για τη δημόσια υγεία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα σε μια προσεχή ευκαιρία να επαληθεύουμε, να ορίσουμε ότι θα επαληθεύουμε και από τα, μας, εθνικά μας συστήματα υγείας ότι ένα φάρμακο το οποίο παίρνει την άδεια και ε, τη σχετική προστασία του, της ευρεσιτεχνίας θα έχει και προσθέμενη αξία. Τη θεραπευτική προσθέμενη αξία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχετε δίκιο που με ευχαριστείτε όντως. Τώρα περνάμε στους αγορητές εξ των πολιτικών ομάδων. Το λόγο για δύο λεπτά έχει η κυρία Αγιούζο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να τονίσω την σημασία της εργασίας της συγκίτριας κύριε Μακάβων, όχι μόνο επί της ουσίας αλλά και επί του τύπου, διότι το έπραξε σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εμπειρογνώμονες των Ισπανικών Αρχών για την βοήθειά τους. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του στήματο προπαγρύπησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, ε, περαιτέρω διεύρυνση της διαφάνειας ε, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το προφίλ ε, κινδύνων που μπορούν να προκαλέσουν κάποια τα φάρμακα αυτά. Θα πρέπει να τονίσουμε την σημασία της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φαρμάκων για την αξιολόγηση που θα κάνει αφορικά με τα προβλήματα ασφάλειας τα οποία ενδέχεται να προκύψουν από τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη την ε, το αποτέλεσμα που είχαμε και η συμφωνία που πετύχαμε σε ζήτημα κοινοποίηση ε, από πλευράς ε, κρατών στις αρμόδιες αρχές. Ε, το Udra Vigilance θα είναι η μοναδική πηγή ενημέρωση, αλλά ταυτόχρονα θα ενημερώνεται και η αρμόδια κρατική αρχή του κράτους μέλους όπου υπάρχει υποψία για ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε τη, σημασία, τη δυνατότητα μάλλον, που δίνεται στους ε, καταναλωτές να μπορούν να αναφέρουν η αδίποτε ε, ανεπιθύμητη ενέργεια και τη δημιουργία μιας ε, ενός πόρταλ ευρωπαϊκού για την συμβολή των πολιτών σε αυτές τις πληροφορίες ε, και την ενημέρωση. Τέτοιο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεδομένου του ότι η φαρμακοπαγρύπνηση διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία της δημόσιας υγείας, η έγκριση της οδηγίας ε, και του σχετικού κανονισμού θα συμβάλλουν σημαντικά στην βελτίωση όχι μόνο των διαδικασιών αλλά και στον συντονισμό των ε, δραστηριοτήτων ανάμεσα στα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη και των αντιστοίχων οργανισμών. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Κορέα Εντεκάμπος έχει το λόγο. Εκ του τη της Ομάδα. Ομάδας. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Η ασφάλεια των νέων φαρμάκων γίνεται γνωστή μόνο αφού κυκλοφορήσουν στην αγορά και αυτό επιβάλλει ένα σύστημα πιο αποτελε... πιο αποτελεσματικό από αυτό που ισχύει τώρα. Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα διαχείρισης κινδύνων αυτή τη στιγμή σε υπερεθνικό επίπεδο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα συστήματα αυτά θα έρχονται πιο κοντά στο πολίτη. Τις τελευταίες δεκαετίες τα φάρμακα έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στον τομέα της δημόσιας υγείας και η ασφαλειά τους και οι παρενέργειες των φαρμάκων Ωστόσο, παρεμένουν ο πέμπτο, η πέμπτη αιτία θανάσου, θανάτου στα νοσοκομεία. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα κοινοτικό σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης βελτιώνοντας τη διαφάνεια και τον συντονισμό. Ο στόχος μας πρέπει να είναι η ε, έγκαιρη ανείχνευση των επιπτώσεων και η αξιολόγηση των παρενεργειών. Τα νέα φάρμακα τα οποία πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης και εποπτείας. Είναι σημαντικό αυτό και πρέπει να γίνουν και ε, μελέτες αποτελεσματικότητας ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις συνέπειες και τις επιπτώσεις αυτών των φαρμάκων στο περιβάλλον. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τη θέση της ΠΡΑΚ και για τις προτάσεις που διατυπώθηκαν. Ευχαριστώ την Ισπανική Προεδρία και την Επιτροπή για τις προσπάθειες και τη συνεργασία τους. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για αυτό το τελικό κείμενο το οποίο θα ψηφιστεί αύριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο για δύο λεπτά, εξ ονόματος των φιλελευθέρων, η κυρία Παρουνάγωβα. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστώ τη Λίντα για την μοναδική ευφία με την οποία χειρίστηκε αυτό το τόσο τεχνικό ζήτημα, καθώ και του σκιώδει συγητές την Επιτροπή και το Συμβούλιο για την επικοδομητική συνεργασία που επεδείχθη τόσο χρήσιμη έτσι ώστε να εξασφαλιστεί αυτή η πρώτη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση για ένα πιο αποτελεσματικό και τυφωνέ σύστημα απεφαρμακοπαγρύπνηση στην, Ευρώ, στην Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν ω και συγκεκριτή από πλευρά τη Άλντα, ε, ιδιαίτερα να ευχαριστώ και την Ισπανική Προεδρία για τι θέσει τη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διατήρησε ε, με επιμονή τι θέσει του κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να πω ότι η φαρμακοεπαγρύπνηση έχει τεράστια σημασία για να εξασφαλιστεί μια σειρά βασικών αρχών που καθοδηγούν τι θέσει τη ομάδα μου και για την εμπιστοσύνη που θα εμπνεύσουμε στον πολίτη αλλά και για την εξασφάλιση υψηλή ποιότητα φαρμάκων. Με τη μέγιστη δυνατή αποδοχή και σε επίπεδο πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με συνεργασία των φαρμακών θρησκευτικών επιχειρήσεων, ε, εταιριών και του κλάδου, του, του κλάδου υγείας. Θα πρέπει λοιπόν να είναι σε θέση οι αρχές να ζητούν μελέτες αποτελεσματικότητας όταν ένα φάρμακο έχει τεθεί στην αγορά και για πρώτη φορά μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία της αξιολόγησης ε, ώστε να μην κινδυνεύει η ζωή του ε, ασθενούς. οι πληροφορίες που θα θα είναι ασφαλείς από καταχρήσεις, αλλά ταυτόχρονα οι ενισχυμένες αυτές τις πληροφορίες που θα συλλέγουμε θα βελτιώσουν την εμπιστοσύνη του πολίτη, του ασθενούς δηλαδή, στην αγωγή που του χορηγείται και θα και ουσιαστικά την ποιότητα των φαρμάκων μας. Έτσι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν την εμπιστοσύνη και κατανόηση του τι είδους φάρμακα είναι αυτά που του έχουν χορηγηθεί. Έτσι μπορούμε να έχουμε μια ευρύτερη ανταγωνιστική και πλήρη αναθεώρηση του φύλου οδηγίων χρήσεως. Έχουμε υψηλή ευθύνη για αποτελεσματικότητα και διαφάνεια ώστε να εξασφαλιστεί ένα καλό σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εξ ονόματος των Πρασίνων. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Τρεμόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την συγγήτρια την κυρία Μακέβαν για το πολύ καλά δουλεμένο σχέδιο έκθεση καθώς και τη συνάδελφό μου στους πράσινους την κυρία ριβασί για την αναλυτική της εργασία. η ανησυχία μας εξ αρχής ήταν ότι στο παρόν σχέδιο υποβόσκει μια τάση να εισάγονται εσπευσμένα φάρμακα στην αγορά χωρίς ενδελεχείς κλινικές δοκιμές και με συνοπτικές διαδικασίες αδειοδότησης με το σκεπτικό ότι θα υπάρχει ένα ενδυναμωμένο σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης ανάλυση κινδύνων και αναφοράς των ανεπιθύμητων παρενεργειών των φαρμάκων. αυτό μας βρήκε αντίθετους εξ αρχή, και σε συνάφεια με τα αιτήματα τη ε, κοινωνίας των πολιτών ζητήσαμε πιο αυστηρές διαδικασίες αδειοδότηση πριν ένα φάρμακο μπει στην αγορά ταυτόχρονα με την παράθεση των αποτελεσμάτων συγκριτικών κλινικών δοκιμών αλλά και την απόδειξη της προστιθέμενης θεραπευτικής του αξίας πιστεύω ότι μέσα από το συμβαστικό κείμενο έγινε προσπάθεια να καμφθεί αυτό το ζήτημα μέσα από την ενδυνάμωση της επιστημονικής επιτροπής φαρμακοεπαγρύπνησης του ευρωπαϊκού οργανισμού φαρμάκων αλλά και την ενδυνάμωση της διαδικασίας αναφορών από τους πολίτες. το δεύτερο που θα ήθελα να σταθώ είναι το θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων των φαρμακευτικών προϊόντων στο οποίο δεν καταφέραμε τελικά μια συμβαστική λύση. η επιτροπή θα έπρεπε μέσω της φαρμακοεπαγρύπνησης να θεσμοθετήσει την υποχρέωση να παρακολουθούνται και να αναφέρονται οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά και να συγκρίνονται αυτά τα δεδομένα με τα αποτελέσματα των δοκιμών που παρουσιάζουν οι εταιρείε κατά τη διαδικασία έγκρισης και διοδότησης των νέων φαρμάκων. δυστυχώς καταφέραμε να έχουμε ε, στο συμβαστικό κείμενο μόνο μια έκκληση στα κράτη μέλη να σκεφτούν το επόμενο στάδιο ε, για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την επιτροπή να παράγει μια αναφορά που θα αναλύει το μέγεθος του προβλήματος και κατά πόσο χρειάζονται τροπολογίες στην υφιστάμενη νομοθεσία. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξ των συντηρητικών για 1,5 λεπτό ο κύριος Καμπνοκ. Ε, Μικρόφωνο σας παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου και εμένα με τη σειρά μου να ευχαριστώ την κυρία Μακάβεν για τη δουλειά που έχει κάνει και όλους ε, όσοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα που συζητούμε. Η οδηγία για τη φαρμακοεπαγρύπνηση έχει παραμείνει απαράλλακτα τα τελευταία δέκα χρόνια. Άρα έχουμε ένα πεδίο περίπλοκο ε, αναθεώρησης και επανεξέταση όλων των θεμάτων μπροστά μας. Πιστεύω ότι η καλύτερη ενημέρωση για τον ασθενή και ισότιμη μεταχείρισή του με τον γιατρό είναι πολύ μεγάλη σημασία. Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης οι διατεθειμένες πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται και στοιχεία σχετικά με ενδεχομένε παρενέργειες των φαρμάκων. η κεντρική βάση δεδομένων που θα συγκεντρώνει αυτά τα στοιχεία, αλλά και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, θα βοηθήσει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος και την αποφυγή μοιραίων πολλές φορές ε, επιπτώσεων. Ε, παραδείγματι, ταχύτατη ε, απόσυρση ενός φαρμάκου από την αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της Ενωτικής Αριστεράς, για δύο λεπτά, ο κ. Μαστάλκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, μιλάμε για ένα σημαντικό θέμα σχετικά με τα φάρμακα. Τα φάρμακα σώζουν ζωές αλλά μπορούν και να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία. Όπως είπαμε προηγουμένως, οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι, ο πέμπτος πιο, είναι το, το πέμπτο πιο σημαντικό ο θανάτου στα νοσοκομεία. Γι' αυτό χρειάζεται ένα διαφανέ και αποτελεσματικό σύστημα φαρμακοεπαγρύπνηση για την ασφάλεια των ασθενών. Με πεπισμένο, Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για αυτό το νομοθετικό κείμενο, καταφέραμε να βελτιώσουμε ουσιαστικά από πλευρά ποιότητα το κείμενο εξασφαλίζοντας καλύτερη προστασία των ασθενών. Συμφωνώ με το σύστημα άμεσης ενημέρωσης, το οποίο μπορούν σε ολόκληρη την Ευρώπη να ενημερώνονται οι ασθενείς για τις παρενέργειες. Οι παρενέργειες μπορούν να εντοπιστούν νωρίς, εφόσον ε, αναφέρονται από τους ασθενείς κάτι που ενδεχομένως θα διστάσουν να συζητήσουν με τον ιατρό τους, αν πρόκειται για παρενέργεια σε ψυχολογικού ή σεξουαλικού χαρακτήρα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης μέσω του διαδικτύου και άλλων μέσων, κάτι πολύ σημαντικό για ασθενείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν οι υπολογιστές. Τονίζεται το δικαίωμα σε ενημέρωση των ασθενών, βελτιώντας την πρόσβασή τους σε πληροφορίες μέσω του ευρωπαϊκού, του ε, ευρωπαϊκού ευρωπαϊκού, της ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης που, υπάρχει, ε, που είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες των κρατών μελών και στη βάση δεδομένων Eurodravigilance. Έχουν λοιπόν σημειωθεί ουσιαστικέ πρόοδοι, αλλά παρόλα τα αυτά το κείμενο χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση. Η διαφάνεια ε, των αρχών λήψη αποφάσεων πρέπει να αυξηθεί. Αυτές οι αρχές πρέπει να καταστούν ανεξάρτητες και ε, βιώσιμες. Επίσης πρέπει να αποφευθεί οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων ώστε να είναι βέβαιο ότι τα μέτρα που θα εφαρμοστούν και θα αποφασιστούν για την προστασία της υγείας των ασθενών δεν θα υπόκεινται σε παρεμβάσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ευχαριστώ κύριο Μαστάλκα. Περνάμε τώρα στους υπόλοιπους αγορητές. Ο κύριο Λίζα έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε. Κυρίε και κύριοι, θέλω να ευχαριστώ ιδιαίτερα την κυρία Μακάβεν, την εισηγήτρια και τους, τη σκιώδη εισηγήτρια από το ΕΛΚ, την κυρία Αϊούσο. Να τι ευχαριστώ ρητά για την δουλειά που κάνανε η κυρία Μακάβεν, αλλά και όλοι οι σκιώδη εισηγητέ έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά, την οποία θα πρέπει να ψηφίσουμε αύριο. Βελτιώνεται σημαντικά η ασφάλεια για τον ασθενή και ε, όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, η μεγαλύτερη πρόοδος είναι ότι χωρίς υπερβολικές αντιπαραθέσεις μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε βελτίωση σημαντική της ενημέρωσης για τον ασθενή. Αυτή η βάση δεδομένου, αυτή η δικτυακή πύλη την οποία θα, έχουν, θα διαθέτουν τα κράτη-μέλη σε κάθε γλώσσα θα βελτιώνει την ενημέρωση του ασθενούς και ταυτόχρονα θα αποτελεί και μια σημαντική ε, βοήθεια για τον ε, ασθενή ο οποίος τη να βρίσκεται σε κάποια ξένη χώρα έτσι ώστε να μην βρίσκεται ανήμπορος ενώπιον ε, στοιχείων άγνωστων που δεν μπορεί να καταλάβει αλλά θα μπορεί μέσα από το ίντερνετ ε, να βλέπει τις πληροφορίες αυτές στη δική του γλώσσα από τη δικτυακή πύλη που έχει προσδοριστεί. Βελτιώνεται λοιπόν και η ενημέρωση πολύ περισσότερο καθώς είναι πολύ καλύτερη από την πρόταση που είχε υποβάλει ο κύριος Φερχόικεν υπό τον τίτλο «Ενημέρωση των ασθενών». Ε, φυσικά θα πρέπει να συμπληρωθεί περαιτέρω το ζήτημα της φαρμακοεπαγρύπνησης, αλλά θεωρώ ότι αποτελεί ήδη η έκθεση και τα όσα έχει κάνει η κυρία Μακέβαν και οι συγκητές ε, πολύ σημαντικά. Κλείνοντας, θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσει το δυνατό η πρόταση για ε, την θέσπιση της, ε, ε, της σχετικής υπηρεσίας, την οποία δυστυχώς μέχρι τώρα έχει η Επιτροπή διαμορφώσει κατά τρόπο ασαφή. Ευχαριστώ. Ε, κύριε, 1,5 λεπτό λόγο κυρία Κάντεμπαχ. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εγώ την κυρία Μαγκέβαν και όλους ε, τους συγητές που συνεργάστηκαν στην υπόθεση αυτή. Θα ήθελα όμως ξεκινώντας να απευθύνω μία έκκληση στους ε, ασθενείς του Ευρωπαϊκού Συστήματος Υγείας. Πιστεύω ότι πρέπει και οφείλουμε και ως ασθενείς ε, και μάλλον σε σχέση με τον ασθενή, ε, να διαθέτουμε επαρκή χρόνο για να, ε, να τον ενημερώνουμε ε, για το τι συνεπάγεται η λήψη ενός φαρμάκου, τι παρενέργειες μπορεί να έχει και ο ασθενής από πλευράς του να δηλώνει, να καταγράφει ό,τι προβλήματα ενδεχομένω συναντήσει. Έτσι μόνο μπορούν να γίνουν τα φάρμακά μας όσο δυνατόν πιο ασφαλή. Βλέπω επίσης ότι οι παρενέργειες καταγράφονται κατά τον ε, τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη που θα επιτρέπει και για το ιατρικό προσωπικό και για τη φαρμακευτική βιομηχανία να ε, ασχοληθούν αμέσω με τι παρενέργειε αυτέ, να τι διαγνώσουν καταρχά, να τι αναγνωρίσουν, να ασχοληθούν με αυτέ και να τι αντιμετωπίσουν. Έτσι μπορούμε να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα, ένα σύστημα που θα λειτουργεί για όλου και ω εκ τούτου μπορώ να χρησιμοποιήσω για το σύστημα της φαρμακοπαγρύπνησης στην Ευρώπη το περίφημο ρητό το όλων σημαίνει περισσότερα και πιστεύω ότι θα πρέπει να εγκριθεί με τη στιγμή την πλειοψηφία η έκθεση αυτή αύριο. Ευχαριστώ κυρία Κάντεμπαχ, κυρία Λεπάζου. το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με τη σειρά μου θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτριά μας την κυρία Μακάβεν για τη δουλειά που έκανε οι συμφωνίες στην πρώτη ανάγνωση δεν ισχύουν πλέον σε αυτό το σώμα διότι μειώνουν τις εξουσίες του Κοινοβουλίου αλλά αυτή είναι ασφαλώς μια πρώτη καλή συμφωνία μετά την πρώτη ανάγνωση. Η κυρία Πανάβανες και η Όδη Συγήτρια έκανε επίσης πάρα πολύ καλή δουλειά. Οι πρόοδοι δεν είναι καθόλου αμελητές, κυρίως ανατομία, ε, το ένα τομέα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη διαφάνεια. Η διαφάνεια πρέπει για μένα είναι ο κανόνας και ο περιορισμός της πρόσβαση στις πληροφορίες να είναι εξαίρεση το μόνο που μπορεί να γίνει αν θέλουμε να έχουμε ε, ολοκληρωμένη ενημέρωση. Η ιδέα να παραμένουν μυστικές οι πληροφορίες που αφορούν την, την, ε, ε, την πνευματική ιδιοκτησία δεν έχουν θέση όταν μιλάμε για την ασφάλεια, την προστασία της υγείας του περιβάλλοντος. Γι' αυτό έχω καταθέσει μια σειρά από τροπολογίες που έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν υψηλό βαθμό διαφάνειας. Θα ήθελα να προχωρήσει περισσότερο, το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε με ικανοποιεί. Το ίδιο το κείμενο, μια διάταξη που είναι σημαντική κατά την άποψή μου, παρόλο που μπορεί να ηχήσει ως ανέκδοτο. Το αίτημα που υποβλήθηκε, που υποβλήθηκε στην Επιτροπή να ελέγξει την ποιότητα των υδάτων και του εδάφους λόγω των καταλήπων των φαρμάκων για να ε, προσδιορίσουμε τις επιπτώσεις της σχετικής νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λεπάζ. Για ένα λεπτό κύριο να έχει το λόγο. Ευχαριστώ η σκιώδηση συγγήτρια δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Μου, μου είπε να σα ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό, για την απουσία τη και να συγχαρώ την κυρία Μακάβαν για το θαυμάσιο τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκε με τι ομάδε για την προετοιμασία αυτού του κειμένου. Το σύστημα τη φαρμακοεπαγρύπνησης των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση είναι κάτι το πολύ σημαντικό και νομίζω ότι καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία θα μα εξασφαλίσει ένα ισχυρότερο σύστημα αξιολόγηση αξιολόγησης κινδύνου, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα χορήγηση αδειών κυκλοφορία και ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο ενημέρωση για οποιοδήποτε παρενέργειε ή ανεπιθύμητε ενέργειε και μεγαλύτερη ασφάλεια των φαρμάκων. Οι ασθενεί θα έχουν καλύτερη πρόσβαση μέσω από δικτυακέ πύλε στην ενημέρωση για πιθανέ παρενέργειε φαρμάκων και τα μέτρα αυτά πιστεύουμε θα ωφελήσουν πάνω απ' όλα του Ευρωπαίου πολίτε και ασθενεί ασθενείς, διευκρινίζοντας και απλοποιώντας το ρόλο της Επιτροπής των κρατών μελών και της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνου και των φαρμακοβιομηχανιών, εξασφαλίζοντας το ψηλότερο βαθμό ασφάλειας. Για τους ασθενείς το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Κάλεμαν. Η κυρία Ματίας έχει λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την οποία επιθυμώ να συγχαρώ στην άμα όλοι γνωρίζουμε πως οι παράπλευρες ενέργειες, οι ανεπιθύμητες ενέργειες συχνά ε, προκαλούν θανάτους ε, στα νοσοκομεία. Για το λόγο. Και τώρα λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε την φάρμακο επαγρύπνηση για φάρμακα τα οποία ήδη κυκλοφορούν ε, στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πλεονέκτημα αυτής της εκθέσεως είναι ότι μέχρι τώρα οι ρυθμίσεις που είχαμε προτείνει δεν κατορθώνουν να ε, λύσουν το πρόβλημα των ανεπιθύμητων ενεργειών. Και αυτό το έχουμε ζήσει με διάφορα φάρμακα, ακόμα και τώρα. Λοιπόν, χρειάζεται να υπάρχει μια εξαντλητική ανάλυση των φαρμάκων. Ε, Θέλουμε λοιπόν ε, μέσω αυτού του συστήματος να καθίσουμε την αγορά πιο διάφανη. Κυρία Γκροστέντε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, μιλάμε για φαρμακοεπεγρύπνηση, σημαντικό πυλώνα του πακέτου φαρμακοεπεγρύπνησης φυτικών προϊόντων, το οποίο δουλεύουμε εδώ και καιρό και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε καλύτερα του ασθενεί απέναντι στου κινδύνου που συνδέονται με τη χρήση φαρμάκων. Αυτή η συμφωνία λοιπόν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ασφάλεια των ασθενών, διότι σπάνια χαρακτηριστικά και σπάνιε ιδιότητε μπορεί να εντοπιστούν έγκαιρα και μια ασφαλή φάρμακα λόγω αυτού θα μπορέσουν γρήγορα να αποσυρθούν από την αγορά αν υπάρχει ανάγκη. Ο σκοπός μας δεν είναι να ξαναδημιουργήσουμε τη φαρμακοπαγρύπνηση, απλώς να βελτιώσουμε την κατάσταση με καλύτερη γνώση των κινδύνων που συνδέονται με τα φάρμακα χάρη σε καλύτερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών. Και η σημασία αυτή τη νομοθεσία αφορά καλύτερη γνώση των ανεπιθύμητων ενεργειών λόγω τη ανάπτυξη τη βάση δεδομένων οργάνων της Vigilance στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων που θα είναι ο μόνος φορέας για την απόξη οποιαδήποτε στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τα φάρμακα. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών. Οι εθνικές αρχές επίσης θα έχουν ευρύτερη δυνατότητα να επαναξιολογήσουν τη σχέση ε, ωφέλους κινδύνου των φαρμάκων ε, αξιοποιώντας όλα τα νέα στοιχεία και ε, ενημερώντας καλύτερα τους επαγγελματίες της υγείας και τους ασθενείς. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν πρέπει να τρομάζουμε τους ασθενείς με προειδοποίησεις οι οποίες θα ήταν υπερβολικές. Θέτοντα τη διάθεση του και ε, αν του παρέχουμε υπερβολικέ πληροφορίε, αυτό μπορεί να αποδειχθεί βλαφερό. Το ένα φάρμακο, ένα σύνθετο προϊόν πρέπει να το εξηγήσουμε με την κατάλληλη ενημέρωση και κυρίω να μην ε, τρομάζουμε υπερβολικά του ασθενεί. Το βλέπουμε αυτό πολύ καλά σήμερα. Σήμερα το, το φύλλο άδεια χρήση έχει χάσει τη σημασία του, είναι δυσανάγνωστο. Πρέπει λοιπόν να το βελτιώσουμε σε συνεργασία με όλου του εταίρου μα, ώστε να υπάρχει από του ασθενεί καλύτερη κατανόηση φαρμάκου και να τους δώσουμε, να τους εμφυσίσουμε νέα εμπιστοσύνη στις ε, επιπτώσεις του φαρμάκου. Ευχαριστώ κυρία Γκροστέτ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Βερνιό έχει το λόγο. Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η φαρμακοεπαγρύπνηση που συνίσταται στην ανάλυση των παρενεργειών του φαρμάκου ε, ώστε ενδεχομένω να αποσυρθούν από την αγορά, από την κυκλοφορία, έχει προκαλέσει λίγο, λίγο ε, ελάχιστο ενδιαφέρον στα πλαίσια τη δέσμη μέτρων για τα φάρμακα. Ωστόσο, είναι κάτι σημαντικό για την ασφάλεια και τη βελτίωση των συστημάτων υγεία μα. Και παρόλο που με χαταχαρά σα βλέπω, κύριε Επίτροπε, λυπάμαι που λείπει σήμερα από την αίθουσα κ. Νταλή, διότι ε, ομολογώ ότι δεν μου άρεσαν καθόλου οι προτάσει επιτροπή οι οποίε έθεταν σε κίνδυνο τη φαρμακοπαγρύπνηση υπέρ των φαρμακοβιομηχανιών. Οι εργασίε του Κοινοβουλίου και του Συμβούλου επέτρεψαν ευτυχώ να βελτιωθεί λιγάκι η κατάσταση. Δεν μπορούμε να γενικεύουμε τι άδειε κυκλοφορία νέων φαρμάκων. Μπορούμε επίση να χαιρετήσουμε τι πρόοδου που έχουν σημειωθεί σε θέματα διαφάνεια. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή είναι μια χαμένη ευκαιρία να βελτιώσουμε τη φαρμακοεπαγρύπνηση και με ανησυχεί η έλλειψη εγγυήσεων για την ανεξαρτησία του συστήματο αν ο ρόλο τη Επιτροπή Αξιολόγηση των Κινδύνων ενισχύεται, δεν, είναι αυτό, δεν παραμένει τελείω ανεξάρτητη ε, από την, Ευρωπαϊκή Επιτροπή που, επιτρέπει την, που χορηγεί την άδεια κυκλοφορία. Αυτή η Επιτροπή έχει κάποιου δισταγμού να επανέλθει στι αποφάσει του. Σε ό,τι αφορά τι εθνικέ δομέ, δεν προβλέπεται για το θέμα αυτό απολύτω τίποτε. Επίση, λυπάμαι που τα κράτη-μέλη δεν χρειάζεται να ανακοινώσουν τυχόν σύγκρουση ενδιαφέρον, συγκρούση ενδιαφέροντο. Και το πιο σοβαρό, αυτή η συμφωνία θέτει τέρμα στην εγγύηση ανεξαρτησία, δηλαδή την δημόσια χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων φαρμακοπαγρύπνους που τώρα πλέον θα χρηματοδοτούνται από ιδιωτικές εισφορές. Ευχαριστώ την Λίντα Μακάβαν η οποία σημείωσε ουσιαστικές πρόοδους σε σχέση με αρχική προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά επειδή υπάρχουν κάποια προβλήματα διαρωτώ με κατά πόσο είναι σκόπιμο να ολοκληρώσουμε μετά από μία ανάγνωση αυτό το φάκελο. Ενώ αν, είχαμε, αν, είχα, το είχαμε εντρυφήσει περισσότερο θα είχαμε πετύχει για τους πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ κυρία Βερνιό. Ένα λεπτό κυρία Ρίσου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η φαρμακοεπαγρύπνηση θα πρέπει να είναι το αντίστοιχο για τα φάρμακα με την αιμοεπαγρύπνηση για το αίμα, δηλαδή να επιτρέπει την αποφυγή κάθε είδους κινδύνου. Το να διαβάσει κανείς και να παρακολουθήσει το φύλλο οδηγιών χρήσεως δεν μπορεί να μας απαλλάξει από κινδύνους όπως εξήγησε η κυρία Μακάβεν ε, υπενθυμίζοντας ε, τις ε, τραγικές περιπτώσεις που γνώρισε η ανθρώπινη ιστορία με φάρμακα που οδήγησαν σε θανάτους ακόμη. Έτσι λοιπόν πρέπει όλοι οι παράγοντες που εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής και κατανάλωσης φαρμάκου να συνεργαστούν με καλύτερο συντονισμό, με ενίσχυση της συνεργασίας και για τον ασθενή, με πληροφορίες δηλαδή οι οποίες θα είναι αμφίδρομες, όπως εξηγήθηκε νωρίτερα, από τους συναδέλφους και με πραγματική διαφάνεια της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης και κλείνω Πρόεδρε. Η ανεξαρτησία των πραγματογνωμόνων αποτελεί το α και το ω κάθε είδους πολιτικής. Εδώ όμως είναι ουσιαδέστα τη σημασία προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του ασθενούς. Για δύο λεπτά το λόγο έχει η κυρία Ευχαρι... Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα να συγχαρώ την κυρία, συγχαρώ την κυρία Μακέβαν και όλους όσους εργάστηκαν ε, στο κείμενο αυτής της οδηγίας τα προβλήματα αυτού του κειμένου είναι πολλαπλά για το σύστημα υγείας και ειδικότερα για την ασφάλεια των ασθενών. Όπως δείχνουν οι στατιστικές, λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών 200.000 άτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο. 50% των ασθενών δεν λαμβάνουν τα φάρμακα σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες και πολλοί ασθενείς θα ήθελαν να έχουν μια αξιόπιστη ενημέρωση με αυτή την ε, αλλαγή στην καταχώρηση των φαρμακευτικών προϊόντων χρειάζεται ένα σύστημα με το οποίο θα μπορούμε μέσω του ίντερνετ να παρέχουμε σωστή ενημέρωση στους διαφερόμενους για τα φάρμακα οι ασθενείς, το, ιατρικό προσωπικό και ε, οι, ε, ε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερώνονται, να ενημερώνονται με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Έτσι, γι' αυτό απαιτείται απόλυτη δημοσιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει σωστά ένα σύστημα φαρμακοπαγρύπνησης με βάση μία ενημέρωση σε όλες τις γλώσσες της κοινότητας ε, μέσω του διαδικτύου το διαδίκτυο είναι μια πολύ χρήσιμη πηγή ενημέρωσης αλλά μπορεί να περιέχει και να μεταφέρει και ασφαλμένες πληροφορίες. Χρειάζεται λοιπόν διαρκής εποπτεία αυτού του συστήματος διότι η αποτελεσματικότητά του έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σε ό,τι αφορά την αυξημένη διαφάνεια του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης γι' αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Πρέπει να συγκεντρώσουμε όλες τις υπάρχουσες πληροφορίες για τις παρενέργειες των φαρμάκων πρέπει να ενημερώσουμε όλα τα μέλη της κοινωνίας και όχι μόνο μια περιορισμένη ομάδα ειδικών για αυτές τις παρενέργειες. Αυτό θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στις φάρμακα. Ευχαριστώ κυρία Λουκατσέσκα. Κυρία Τσίλντερ, έχει το λόγο. Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφη κυρία Μακάβαν για την έκθεσή της. 200.000 θάνατοι όμως το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφειλόμενοι σε παρενέργειες από φάρμακα που έχουν στακρογραφηθεί, σημαίνουν ότι χρειάζεται πράγματι ένα σύστημα που θα παρακολουθεί την ασφάλεια των φαρμάκων, ακόμη και μετά την έγκρισή τους. Οι παρενέργειες αποτελούν την πέμπτη σε σειρά αιτία ε, νοσηλεία σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία. Έτσι λοιπόν μετά την αδειοδότηση και διάθεση στην αγορά των φαρμάκων πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση σε συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών που θα παρακολουθούν και τον κίνδυνο να διατεθούν στην αγορά παραποιημένα ή αλλοιωμένα φάρμακα που αποτελούν απελπίσει πολύ μεγάλο κίνδυνο σήμερα. Η αλλοιωμενα φαρμακα που αποτελουν να περιπισει μέσα από το φύλλο οδηγιών χρήσεως για τον ασθενή θα βελτιώσουν ασφαλώς την υγεία και την ασφάλεια για όλους τους πολίτες στην Ευρώπη. Η ε, δικτυακή πύλη που θα θεσπιστεί σε κάθε χώρα και σε κάθε γλώσσα θα επιτρέπουν επίσης ε, στους ασθενείς να βρίσκουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά ο κύριος Μπαρτολότσι. Ναι, πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Ναι, αυτό το νομοθέτημα θέλουμε να ορθολογικοποιήσουμε το σύστημα της ευρωφύλαξης της ε, στην Ευρώπη. Οι προτάσεις της ε, κυρίας Μακέβα τροποποιούν τον κανονισμό 726 αλλά και την οδηγία 83 του 2001. Χάρη λοιπόν στην αγαστή συνεργασία Κοινοβουλίου Συμβουλίου αλλά και των συναρμοδίων κοινοβουλευτικών επιτροπών μπορέσαμε να καταλήξουμε στο να συζητάμε σήμερα μια πρόταση που αστοχεύει στοχεύει στη βελτίωση του συστήματος της φάρμακοπαγρύπνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην τελειοποίηση των δραστηριοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον τομέα απλούστευση, διαφάνεια και ορθολογικοποίηση μπορούν να θεωρηθούν ως τα σημεία κλειδιά αυτές της ε, έκθεσης που προτείνουν μέτρα που στοχεύουν στην ε, καλύτερη προστασία της ε, ανθρώπινης υγείας και με εναρμονισμένο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια να γίνονται αναφορά σε μέσα τα οποία αφορούν τόσο την τον καθορισμό των ρόλων των εμπλεκομένων τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο αλλά και σε μια πιο ενεργό ε, συμμετοχή του ασθενούς στον οποίο αναγνωρίζεται θεμελιώδης ρόλος για την ενίσχυση της διαφάνειας, της πληροφόρησης ε, σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων αλλά και περαιτέρω στην απλούστευση της αξιολόγησης, ενημέρωσης σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Ε, το σύστημα της φαρμακοπαχνύπνησης θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω χάρη στην πιο στενή συνεργασία σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μια αποτελεσματική συμμετοχή και στα τρία 7 επίπεδα θα εγγυηθεί μια σωστή ανταλλαγή προφοριών που θα αφορούν τις παρενέργειες των φαρμάκων. Το νέο σύστημα της φαρμακοεπαγρύπνησης θα πρέπει να οργανωθεί ως δίκτυο και μέσω της χρήσης του διαδικτύου και να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο ενημέρωσης, ενημέρωσης ασφαλούς με συμμετοχή των εμπλεκομένων ε, ευχαριστώ κύριε Μπαρτολότσι. Για δύο λεπτά το λόγο κύριος Μαρινέσκου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο τομέας αυτός είναι ένας ε, τομέας πολύ σημαντικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση που οφείλεται στην άμεση σχέση που έχει με την ε, ασφάλεια η οδηγία και ο κανονισμό τον οποίο συζητάμε σήμερα θα επιτρέψει τη βελτίωση του συστήματο φαρμακαγρύπνηση. Προβλέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στι εθνικέ και τι ευρωπαϊκέ αρχέ και μια συνεχή επαφή με του εκπροσώπου τη βιομηχανία αλλά και των ασθενών τα στοιχεία σχετικά με τις ανεπιθύμητες ε, ενέργειες των φαρμάκων θα είναι προσβάσιμο τόσο στους επαγγελματίες του κλάδου όσο και στις αρμόδιες αρχές αλλά θα είναι και διαθέσιμο στους ασθενείς, στους πολίτες που θα πρέπει να γνωρίζουν όλα τα χαρακτηριστικά των φαρμάκων που χρησιμοποιούν και αυτή η πληροφορία θα πρέπει να αναφέρεται ε, ρητά στο φύλλο χρήσης, φύλλο μάλλον του φάρμακος. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε εποχέ όπου δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε τι ανεπιθύμητε ενέργειε των φαρμάκων, ενώ τώρα μπορούν να εντοπιστούν πολύ καλύτερα χάρη στο νέο σύστημα. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε μια φάρμακαπρίμπηση επαρκώ ε, ρυθμιζόμενη και να υπάρχει ενημέρωση ανά πενταετία. Οι ανεπιθύμητε ενέργειες των φαρμάκων μπορούν να ε, εντοπιστούν ακόμα και αν έχουν ε, παρέλθει 30 χρόνια από την αδειοδότηση του φάρμακου. Θα πρέπει επίσης να αναφερθούμε στην αλληλεξάρτηση που υπάρχει ε, ανάμεσα στον φαρμακευτικό κλάδο και τις, και τεχνολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαρουνέσκου. Για δύο λεπτά το λόγο έχει η κυρία Ροντζούλη. Κύριε Πρόεδρε, Πίτρο Πεταγιάννη, η επαλήθευση της ασφάλειας των φαρμάκων αφού αδειοδοτηθούν είναι το βασικό στοιχείο αυτής της πρώτης κανονισμού. Οι αξιολογήσεις και οι ε, θετικές ή αρνητικές δεν είναι ποτέ υπερβολικές. Το θέμα ότι το ζήτημα ότι 55 θάνατοι ετησίως οφείλονται στα φάρμακα είναι πολύ σοβαρό. Συχνά αυτές οι, αυτοί οι έλεγχοι, αν γίνονται σε τακτά διαστήματα, μπορούν να εντοπίσουν αυτές τις ε, παρενέργειες, που μπορεί να οφείλονται και σε ε, χρήση, συνδυασμό μάλλον ε, διαφόρων φαρμάκων. Θα πρέπει λοιπόν η φαρμακοπαγρύπνηση να είναι μία από τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα καλό σύστημα φαρμακοπαγρύπνησης θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτρέπει στους, ε, σε υπηρεσίε και στους ασθενείς να σημειώνουν τις διάφορες αρνητικές επιπτώσεις, ανεπιθύμιες συνέργειες ε, κλπ. Μόλις ε, εντοπιστούν λοιπόν αυτά τα μηνύματα θα πρέπει να δράσουμε π.χ. τροποποιώντας τον τρόπο με τον οποίο χορηγείται ένα φάρμακο, βελτιώνοντας την χρήση του, αλλά και ενδεχόμενα την, την απόσυρση του φάρμακου σε, σε περιπτώσεις σοβαρών ε, ανεπιθύμητων ενεργειών. Η συνεργασία λοιπόν ανάμεσα στους εμπλεκομένους τομείς θα έχει θετικά αποτελέσματα διότι θα μπορούμε έτσι να ελέγχουμε περισσότερο τους ε, ανοιχνεύσεις οι οποίες θα γίνονται και έτσι θα μπορούμε να αποσύρουμε τάχιστα από την κυκλοφορία ε, συσκευάσματα τα οποία είναι επικίνδυνα. Όλα τα κράτη-μέλη θα συνεχίσει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της φαρμακαγρύπνησης και κατά λίγο πρόεδρε τονίζοντας ε, τη σημασία που έχει η άμεση συμμετοχή των ασθενών στην, ε, και τις αυθόρμητες αναφορές που γίνονται από ε, τους ασθενείς σε εθνικές αρμόδιες αρχές. Θα πρέπει να τονίσω ότι στις χώρες όπου αυτό εφαρμόζεται δεν επιφέρει κανέναν επιπλέον άχρος ε, από τις αρμόδιες αρχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ροντσούλη. Και τώρα περνάμε στο Catch the Eye. Για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Κορκουνέντε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η πιο σημαντική πτυχή, πιστεύω, στο έγγραφο είναι καταρχάς η βάση δεδομένων και ε, οι πληροφορίες που διατίθεται. από ένα κεντρικό σημείο σε όλους τους ασθενείς. Από εκατοντάδες από 200.000 θανάτους που έχουμε θα μπορούσαμε να μειώσουμε σημαντικά τον αριθμό έχοντας, ε, στη διάθεση, προσφέροντας τη διάθεση του ασθενούς απλώς και μόνο καλές πληροφορίες για παρενέργειες. Και βλέπουμε ότι ανάλογα με τη χώρα υπάρχουν και διαφορετικά ε, ποσοστά. Πολλές φορές δε η διαφορά στα αριθμητικά στοιχεία, δηλαδή στα ποσοστά θανάτων που διαπιστώνονται από ότι μια χώρα στην άλλη, έχει να κάνει και ή κυρίως με την ελληπή ενημέρωση από τον θεράποντα ιατρό προς τον ασθενή. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι η ενημέρωση θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επίσης, η ενημέρωση για τις παρενέργειες πρέπει να έρχεται εγκαίρως και όχι με καθυστέρηση. Ιδιαίτερο ρόλο φυσικά έχουν να διαδραματίσουν και οι αρμόδιε αρχέ. Οι ευθύνε μα είναι πολύ μεγάλε. Ευχαριστώ, κύριε Νικολάσου. Ευχαριστώ το Πρόεδρε. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ενημερώνουν όχι μόνο τις σοβαρές, αλλά όλες τις περιπτώσεις στη βάση δεδομένων της φαρμακοεπαγρύπνησης, ώστε όλα τα στοιχεία να συγκεντρώνονται σε έναν ενιαίο χώρο, σε αυτή τη βάση που θα αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την έρευνα. Έτσι θα μπορούν να ληφθούν μέτρα για την αλλαγή του τρόπου συνταγογράφησης, για την καλύτερη ενημέρωση των ασθενών για το φάρμακα και για την απόσυρσή του από την αγορά. Υποστηρίζουμε τα μέτρα που έχουν σκοπό να ενθαρρύνουν τους ασθενείς να ενημερώνονται, να γνωρίζουν όλες τις πληροφορίες για το φάρμακο διαβάζοντας τις οδηγίες χρήσης. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο θα γνωρίζουν ποιες είναι οι τυχόν παρενέργειες του φαρμάκου, αλλά θα μπορούν να γνωρίζουν όπως είπαμε τις παρενέργειες και αυτές οι παρενέργειες να είναι γνωστές σε όλους. Η έκθεση της κυρίας Μακέβαν αποτελεί μια ουσιαστική πρόοδο υπέρ της ασφάλειας και της ενημέρωσης των ασθενών στην Ευρώπη. Κυρία Βάισμπεργκερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την καταπληκτική της δουλειά και, ε, την, ε, και θα ήθελα να πω ότι η καλή φαρμακοεπραγρήμηση προστατεύει τον πολίτη και ενθαρρύνει τον ασθενή στη χρήση των φαρμάκων που χρειάζεται να λάβει. Είναι πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν οι δικτυακέ πύλε για του ασθενεί, η ενημέρωση, η συλλογή των στοιχείων. Θετικό στοιχείο είναι επίση ότι αύριο θα έχουμε δικτυακές πύλες με καλή ενημέρωση, με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο ασθενής. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν θέτουμε ένα τέρμα σε μία ε, απαράδεκτη κατάσταση, γιατί μέχρι τώρα σε ορισμένα κρατημέλη δεν ήταν υποχρεωτική η δημοσίευση του φύλου οδηγιών χρήσεως στο διαδίκτυο. Μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε αυτή την ενημέρωση έχοντας στην διάθεση του ασθενούς το φύλλο διγιών χρήσεων στη γλώσσα του, αλλά επίσης και στο διαδίκτυο διαθέσιμο, έτσι ώστε αν κάνει το χάσει ή δεν έχει τον τρόπο να το ξαναβρει, να μπορεί να το αναζητήσει από το διαδίκτυο. Και θα ήθελα να παρακαλέσω να γίνουν δεκτές οι τροπολογίες. Μας ευχαριστώ πολύ την κυρία Βάισπερ και Το λόγο έχει η κυρία Ριβασί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στις περιβαλλοντικές συνέπειες που έχουν τα φάρμακα από το 65 και μετά η Ευρώπη κατέρτισε κριτήρια για την αδειοδότηση, για διάθεση στην αγορά που βασίζεται σε τρία κριτήρια. Η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και η φαρμακευτική ποιότητα του φαρμάκου, αλλά τίποτα στον αφορά τον αντίκτυπο που έχουν τα φάρμακα στο περιβάλλον. Αλλά θα ξέρετε ότι επί του παρόντος ότι τα ιστρογόνα που βρίσκονται στα περιοχές των ποταμών αλλάζει το φύλλο των ψαριών. Γνωρίζετε ότι βρίσκουμε κατάλοιπα και στους σταθμούς καθαρισμού και στα απόβλητα των νοσοκομείων ε, που δείχνει πόσο σημαντικά είναι τα κατάλοιπα των φαρμάκων. Διεξήχθη μια συζήτηση, συζητήθηκε αρκετά και όσον αφορά την την σχετική οδηγία, ε, λήφθησαν υπόψη αυτά σε αιτιολογικές σκέψεις που ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συναρτήσει των δεδομένων που δίνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων, η Υπηρεσία για το Περιβάλλον και τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύει μια έκθεση όσον αφορά το εύρο του προβλήματο και μια αξιολόγηση όσον αφορά την ανάγκη και χρησιμότητα να τροποποιηθεί η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω όσον αφορά τα φάρμακα σε διάφορου τομεί. Και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα πει θα ετοιμάσει μια έκθεση βάσει αυτών των δεδομένων, διότι έμεσα τελικά αυτό επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία, διότι υπήρχαν πολλές περιπτώσεις που μέσω, ε, είχαμε δευτερεύουσε συνέπειε μέσω κατανάλωση υδάτο. Ευχαριστώ για ένα λεπτό. Ο κύριο Ντόρφμαν έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ισηγητά, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι συζητούμε σήμερα για το ζήτημα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να θίξω ένα ζήτημα το οποίο είναι σημαντικό για μένα. Είναι η πολυγλωσία στην πληροφορία που περιέχεται στα, στα φάρμακα αυτά. Ε, δεν πρόκειται μονάχα για μειονοτικές γλώσσες. Πολλές φορές είναι πρόβλημα σε περιοχές που υπάρχει μεγάλη τουριστική ροή. Στη δική μου περιοχή, παραγματικά υπάρχει ένα μεγάλο μέρος με ανθρώπων οι οποίοι δεν κατανοούν τις οδηγίες οι οποίες βρίσκονται στα φάρμακα. Αυτό δεν είναι μονάχα δυσάρεστο, είναι και επικίνδυνο. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε στο τομέα αυτό και να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες είναι δυνατόν να είναι ανακτήσιμες από το διαδίκτυο για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν αυτά που λένε τα φάρμακα σε ένα συγκεκριμένο χώρο και αυτές οι πληροφορίες επίσης να είναι σε μια μορφή εύληπτη και συνοπτική ώστε να μπορούν να κατανοούν οι πολίτες περί τίνος πρόκειται και να υπάρχει μια, μια σύντομη σύνοψή τους στα στα φυλάδια τα οποία συνοδεύουν τα φάκελ, τους, ε, του, τα φάρμακα ώστε να μπορούν να κατανοούν περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστώ πολύ λέει και ο Πρόεδρος. Ο κύριος Ρώση για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε υπέρ τη τοποθετήσεω τη συγγήτρια που τονίζει τη σημασία που έχει να επαλέξουμε κατά πόσο είναι ασφαλή τα φάρμακα και να βελτιώσουμε τη διαφάνεια όσον αφορά ε, την φαρμακοεπαγρύπνηση. Η Λέγα του Βορρά υπογραμμίζει και υπογράμμισε κάποιε στοιχεία. Να επιτρέψουμε την άμεση πρόσβαση των ασθενών στη Τράπεζα Δεδομένων την κοινοτική όσον αφορά τι ύποπτε αντιδράσει ε, θα πρέπει να υπάρχουν διάφορες ε, τιμολογήσει των κατών μελών που θα αξιολογούν και στην ε, αποτίμηση που γίνεται μέσω της φαρμακοπαχρύπνησης και θα πρέπει να δοθεί και στην, ε, στην Επιτροπή την αρμόδια για την αξιολόγηση των κινδύνων. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ε, κρίσης και τα κράτη-μέλη και οι φορείς και οι ασθενείς. Λοιπόν, είναι, είναι, επιβάλλονται φάρμακα με αρνητικέ συνέπειε ενδεχόμενε ε, και φυτογενεμικά φάρμακα, διάφορα φάρμακα. Και γι' αυτό μπορεί ευαίσθητοι να έχουν απολεργικέ αντιδράσει μέχρι να αποστούν οι σοβαρέ ασθένειε που είναι ει βάρος των ανθρώπων. Ε, κάτι που δεν είναι κάτι γνωστό μέχρι σήμερα και που δυστυχώ δεν είναι εύκολο να επιληθεί το πρόβλημα είναι το πολλαπλό χημικό σύνδρομο. Όποιο πληγεί από αυτό δεν μπορεί να ζήσει κανονική ζωή, διότι δεν ανέχεται την επαφή με κανένα χημικό προϊόν. Είναι λοιπόν σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να δραστηριοποιηθεί ούτω ώστε να ενημερώσει και να καταρτήσει του πολίτε για την ε, σοβαρή επίγνωση με γνώση χρήση των φαρμάκων. Ευχαριστώ κύριε Ρώση. Ο κύριος Σνέρχαρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Αν σκεφτεί κανείς πώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας θητείας ξεκινήσαμε να συζητούμε για την προβληματική του θέματος αυτού, μπορεί να έχει μόνο σεβασμό και δέος ενώπιον του εισηγητού που κατάφερε να φέρει αυτό το θέμα σε περαίωση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η φαρμακοεπαγρύπνηση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη είναι εντυπωσιακό ότι τελικά αποδέχτηκαν να υπάρξει μια τράπεζα δεδομένων η οποία να έχει διασύνδεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θέλουμε επίσης να ζητήσουμε από την Κομισιόν να υπάρξουν οι απαραίτητες δυνατότητες να χρησιμοποιούν οι διάφοροι φορείς της Κομισιόν τις τράπεζες δεδομένων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που θα τη βοηθήσει να κατανοήσει την κατάσταση των φαρμάκων και να υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη της ποιότητός τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πάρα πολλοί πολίτες αναφέρουν ότι είναι απαραίτητο να έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα με παρενέργειε και επομένω είναι απαραίτητο να υπάρχει η σωστή τεκμηρίωση για όλα τα σκευάσματα ώστε να αποφεύγονται στο βαθμό του δυνατού οι παρενέργειε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Ρίκε έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Μια σύντομη παρέμβαση. Θέλω να συγχαρώ όλου εκείνου που επεξεργάστηκαν το θέμα και με εκπλήσει ένα σημείο το οποίο δεν εκαλύφθη. Η ήτη φαρμακοπεγρύπνηση, διασταυρούμενη φαρμακοπεγρύπνηση κάθετα στα κάθετα, σε κάθε προσέγγιση των προϊόντων εξαντλητική η έκθεση, όμως οι περισσότερα, περισσότερα προβλήματα προέρχονται από το 182% ε, παίρνουν πάρα πολλά φάρμακα παράλληλα οι, οι ασθενείς και μπορεί ένα φάρμακο κάθετα να μην έχει ιδιαίτερε συνέπειε, να έχει δευτερεύουσες τοξικές συνέπειε αν διασταυρούνται με ένα άλλο φάρμακο. Είναι ύψη τη σημασία λοιπόν να μπορέσουμε να έχουμε μια βάση δεδομένων όσον αφορά τι συνέπειε δεσταυρούμενε των φαρμάκων που θα είναι στη διάθεση και των επαγγελματιών και των ασθενών. Και αυτό είναι ακόμα πιο αναγκαίο διότι πάρα πολλοί ασθενεί ε, έχουν κατόπιν συνταγή, ε, έχουν συνταγολόγιο, παίρνουν φάρμακα με συνταγή και παίρνουν και άλλα φάρμακα. Και δεν υπάρχουν ενδείξει όσον αφορά τι ε, τοξικέ συνέπειε διασταυρώσεω φαρμάκων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ακροθυγώ εξετάστηκε και είναι πάρα πολύ λυπηρό κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρος, κύριε Ρίκε. Δίνω τώρα το λόγο στο Συμβούλιο, στον Υφυπουργό κύριο Σαστέαο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, απλώς θέλω να αναφέρω με λίγα λόγια τις ευχαριστίες μου και τα συγχαρητήριά μου στην κυρία Μακάβαν, και τους ε, συζητητέ, όπω βέβαια και την Κομισιόν και την Ισπανική Προεδρία για το έργο το οποίο επετέλεσαν να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο είναι ισορροπημένο μένα αλλά και πάρα πολύ ζωτικό για το σύνολο των ασθενών σε ευρωπαϊκό έδαφο. Αυτό το θέμα είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα τη προσθέμενης αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη ζωή των συμπολιτών μα και τη εφαρμογή. η εφαρμογή μάλλον αυτή, αυτών των ρητρών θα επιτρέψει να μειωθούν σημαντικά οι περιπτώσεις όπου έχουν παρουσιαστεί παρενέργειες ανεπιθύμητες από την χρήση φαρμακευτικών συσκευασμάτων, που όπως ξέρετε είναι και ένας από τους βασικούς λόγους θνησιμότητος στα νοσοκομεία. Γι' αυτό λοιπόν εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι σε πρώτη ανάγνωση τίθενται ε, σε ψηφοφορία όλοι αυτοί οι σαφείς και αποτελεσματικοί κανόνες φαρμακοεπαγρύπνησης. Ελπίζω ότι μέχρι το τέλος της Βελγικής Προεδρίας θα μπορέσουμε να έχουμε και πρόοδο στα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Ήδη το Συμβούλιο μαζί με την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο θέλει να προωθήσει όλα αυτά τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τόσο πολύ του Ευρωπαίου πολίτε και ιδίω του ασθενεί στον φαρμακευτικό τομέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρο. Δίνω τώρα το λόγο στον Επίτροπο Ταγιάννη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι η συζήτηση που έλαβε χώρα σήμερα με τη συμμετοχή πολλών βουλευτών δείχνει τη σημασία που έχει η συμφωνία η οποία πετεύχθη μεταξύ των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Ισχυρό μήνυμα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στέλνουν προς τους πολίτες της Ένωσής μας, της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης, που είναι κάτι που θα ενισχυθεί και από τα χαρτοφυλάκια που θα εγκριθούν γρήγορα, ελπίζω, όσον αφορά τα περιμένα χράματα, τις πληροφορίες που πρέπει να δίνονται στους ασθενείς και συμμερίζομαι μάλιστα και τις ανησυχίες που εξεφράστησαν κατά τη διάρκεια της συζητήσεων αφορά τους θανάτους που προξενήθηκαν από φάρμακα που δεν εσεβόνταν τις προδιαγραφές. Κάτι που αναφέρθηκε και η κυρία Νούτη ήρθε και με το νεογέννητο παιδί της εδώ. Ευτυχώς αυξάνεται να μεγαλώνουν με ευρωπαϊστικά συναισθήματα τα παιδιά. Και αυτά που είπε ο κ. Ντόφμαν, ο καθένας από εμά πράγματι μπορεί να εκφραστεί στην γλώσσα του και μπορεί να γνωρίζει στην μητρική του γλώσσα τις ε, προδιαγραφές που ε, εγγυώνται την ασφάλεια όσον αφορά τη χρήση των φαρμάκων. Εγώ υποστηρίζω την πολυγλωσία σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα με τον οποίο ασχολούμαι κανονικά. Θα ήθελα να καθησυχάσω και κύριο Βερνιό για τις ε, ανησυχίες που εκφράστηκαν. Ευχαριστώ εν ονόματι ως Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν και ο Επιτροπός Ντάλι δεν ήρθε σήμερα αλλά θα ενημερωθεί για την συζήτηση και θα του διαβιβάσω όλες τις παρατηρήσεις που έκαναν όλοι οι αξιότιμοι βουλευτές οι οποίοι συμμετείχαν στην σημερινή συνεδρίαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας ευχαριστά εκ βάθους καρδίας διότι μπορεί δώσαμε ένα ισχυρό μήνυμα προς συμπολίτε της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όσον αφορά τώρα το θέμα που έθεσε η κυρία Ριβάση, όσον αφορά την ενίσχυση των κανόνων σχετικά με, τον, με τους κινδύνους που δημιουργούν τα φάρμακα στο περιβάλλον, πρέπει να πούμε ότι εκτιμούμε και εμείς το σημαντικό να ληφθούν πτυχέ προστασία του περιβάλλοντο και δεχόμαστε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που να υποβληθεί μια έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, που θα συνοδεύεται ενδεχομένω από νομοθετική πρόταση σχετικά με του κινδύνου που δημιουργούν τα φάρμακα στο περιβάλλον. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου προσφέρετε έτσι για να επενθυμίσω στι κυρίε και κυρίου βουλευτέ ότι οι περιβαλλοντικέ πτυχέ ήδη σε σαν σημείο δράση στην ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούσε το μέλλον του φαρμακευτικού τομέα και ε, θα υιοθετηθεί στο, θα, που παρουσιάστηκε μάλλον ήταν και διάφορα μέτρα που θετήθηκαν στο πακέτο που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2008 για τα φάρμακα. Ευχαριστώ Επίτροπε. Θέλει και η Προεδρία της Συνόδου να ευχαριστήσει και την κυρία Τσούλη για τον τρόπο με τον οποίο έχει συνδυάσει εντυπωσιακά την οικογενειακή ζωή και την εργασία. Κύριε Αντσούλη, σας θαυμάζουμε όλοι. Έχει το λόγο τώρα η συγγήτρια κυρία Μακάβαν για να κλείσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω σε κάποια από τα σημεία που πεθύγησαν. Μίλησαν συνάδελφοι για διαφάνεια. Θα ήθελα να πω ότι αυτό που πετύχαμε είναι μεγάλο βήμα προόδου για τη διαφάνεια. Οι πληροφορίε που θα δίδονται δημόσια μέσω των διαφόρων ε, ιστοτόπων είναι τεράστια αύξηση σε σχέση με τα ήδη χορηγούμενα. Και όσον αφορά την αναξαρτησία του έργου τη φαρμακοεπαγρύπνηση, αυτό φαίνονταν σε δουλειά που έκανε το Κοινοβούλιο, που την αδειοδότηση τη διαχώρισε από την φαρμακοεπαγρύπνηση. Αν η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνηση κάνει συστάσει, οι συστάσει θα ανατρέπονται μόνο αν υπάρχουν άλλε αποδείξει. Κάναμε σημαντική προσπάθεια να βελτιώσουμε την ανεξαρτησία του φορέα. Επίτροπε, πολλή δουλειά πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από την έγκριση τη νομοθεσία αύριο. Νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο που την εγκρίνει. Πολλή δουλειά πρέπει να γίνει για το φυλάδιο ενημέρωση των ασθενών. Πολύ δυσαρέσκεια εκφράζεται από οργανώσει ασθενών και από ασθενεί μεμονωμένου περί αυτό. Εσεί προσπαθήσατε να βρείτε μια λύση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ήταν αυτή που θα γινόταν αποδεκτή, αλλά θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σα, ώστε να έχουμε ένα καλό φυλάδιο για την ενημέρωση του φυλάδιο δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει τα πάντα που μπορούν να συμβούν σε έναν ασθενή, διότι τότε θα ήταν άχρηστο το φυλάδιο για τον μέσο ασθενή. Θα πρέπει να είναι κάτι λογικό, θα πρέπει να παρέχει πληροφορίε, πρέπει να συνεργαστούμε από αυτού. Θα ετοιμάσετε την μελέτη όσον αφορά τι ε, περιβαλλοντικέ συνέπειε που έχουν τα φάρμακα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλουμε να δούμε και το μαύρο σύμβολο. Θέλουμε αυτό το σύμβολο να αναπτυχθεί, δεν θέλουμε να απομακρυνθεί όπως, κάναμε, όπως συνέβη όσον αφορά τα φάρμακα για τα παιδιά, τα παιδιατρικά φάρμακα. Θέλουμε αυτό το σύμβολο σύντομα να εμφανιστεί. Τώρα όσον αφορά τα κράτη-μέλη πρέπει να γίνει πάρα πολύ δουλειά όσον αφορά τις, τους διάφορους ιστοτόπους. Θέλουμε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Είναι σημαντικό κόσμος να παίρνει στη γλώσσα του πληροφορίες και τα κράτη-μέλη επίσης θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα σύστημα άμεσης ενημέρωσης. Αυτό φορά πολλούς εθνικούς φορείς. Όσον αφορά την ΕΜΑ, ε, την ΕΜΕΑ πρέπει να γίνει πολλή δουλειά, χρειάζονται σωστοί πόροι και το συζητούμε αυτό και το συζητήσαμε με μακρόν στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστούμε όλους τους ενδιαφερόμενους, ελπίζουμε να είναι μεγάλη πλειοψηφία αύριο και τότε η πραγματική δουλειά μπορεί να ξεκινήσει ούτως ώστε να κάνουμε τη διαφορά επιτόπου για τη ζωή των ανθρώπων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κλείνει η συζήτηση λοιπόν για το σημείο αυτό τη σημερινής της Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο τη σημερινής της είναι η έκθεση της κυρία Κλάς σε σχέση με την ε, εμπορία και την χρήση βιο